Ω δημοκράτη, πρέπει να πω όχι και γι' αυτό θα πούμε όχι σε αυτές τις εκθέσει αύριο. Σας ευχαριστώ κύριε Έρλα για τους μη εγγεγραμμένου. η κυρία Στάσεν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε.